Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ μέσα όπως βλέπετε έχει γίνει μια επανάσταση. Ο πρόεδρος και πολλοί αντιπρόεδροι εξαφανίστηκαν. Όχι γιατί φοβήθηκαν τους αστυνομικούς που ήρθαν εδώ, αλλά για άλλους λόγους, άγνωστους. Και ο μόνος ευρωβουλευτής εδώ είμαι εγώ, άρα δεν μπορούσα παρά να προεδρεύσω θα συζητήσουμε όλοι μαζί το θέμα του οργανωμένου διεθνούς εγκαλήματος και την αξιολόγηση της απειλής που αντιπροσωπεύει το μεγάλο οργανωμένο έγκλημα. Αρχίζει τώρα ένας καινούργιος κύκλος, 13 με 17. Η Ευρωπόλ μόλις δημοσίευσε μία αξιολόγηση της απειλής από το οργανωμένο έγκλημα και υπάρχουν και επισκέπτες από την Επιτροπή Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επίσκεψή τους ίσως δείχνει ότι μπορεί να θελήσουν να παραμείνουν στην Ένωση. Τέλος πάντων τελείωσαν τα αστεία τώρα. Τώρα τα σοβαρά. Η συμβολή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή ποια είναι. Θα ακούσουμε τον Διευθυντή της Ευρωπόλ, τον κύριο Γουέιν Ράιτ, για περίπου 15 λεπτά και μετά θα ακούσουμε τον Μάρτιν Πάουερ, πρόεδρο της Κόζη, για άλλα 15 λεπτά. Και μετά θα δούμε αν είναι κανείς σε θέση να σχολιάσει. Μετά όμως αυτά μετά. Ορίστε κύριε Wainwright μου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Παρά την φαινόμενη έλλειψη ενδιαφέροντος στην Επιτροπή σας, χαίρομαι για την παρουσία μου εδώ, όπου θα παρουσιάσω τα συμπεράσματα της αξιολόγησης μας, της τελευταίας μας αξιολόγησης που είναι η πιο λεπτομερής που έχει ποτέ γίνει. Για πρώτη μάλιστα φορά πήρε στοιχεία ευρύτερα από ακαδημαϊκούς για να είμαστε βέβαιοι ότι η μεθοδολογία που θα ακολουθούσαμε θα ήταν η καταλληλότερη. Κάνουμε πολλές αξιολογίες στην Ευρωπόλ, αλλά αυτό είναι το κυριότερο προϊόν μας. Μαζεύαμε στοιχεία επί δύο χρόνια ολόκληρα και Βασίζεται η μελέτη αυτή στις τελευταίες αποφάσεις της Ένωσης για την αντιμετώπιση του ενωμένου κλίματος. Βλέπετε και από τις διαφάνειες αλλά και από τη δημοσίευση που κάναμε αυτή την εβδομάδα ότι κάναμε και ορισμένε συστάσεις για τις πιο σημαντικές απειλές που θα αντιμετωπίσουμε ως οργανωμένο έγκλημα. Το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης σε λίγες εβδομάδες θα θελήσει να καθορίσει στρατηγικές προτεραιότητες για τα επόμενα τέσσερα χρόνια στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ένωση, στην Ευρωπαϊκή μάλιστα Ένωση. Τώρα, πώς καταλήξαμε σε αυτά τα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Στην αξιολόγηση μας συμπεριλάβαμε κρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται όλο και πιο δυναμικό και πολύπλοκο το οργανωμένο έγκλημα και το οποίο παραμένει σημαντική απειλή στην ευημερία της Ένωσης. Παρατηρήσαμε παραδείγματο χάρη από τότε που ξέσπασε η οικονομική κρίση ότι αυξήθηκε η μαύρη αγορά και η σκιώδης οικονομία με παράνομα κέρδη δισεκατομμυρίων πράγμα το οποίο πλήττει και τις δυνατότητές μας να βγούμε από την κρίση. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οργανωμένων κλίματος στην ενωση 500.600 περίπου. Η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει και καινούργιες νέες παραλλαγές της εγκληματικής δραστηριότητας και οι παραδοσιακές βέβαια δραστηριότητες όπως το λαθρεμπόριο ναρκωτικών αλλά και καινούργιε δυνατότητες κατάχρησης και εκμετάλλευσης της νομοθεσίας για εγκληματικά και παράνομα κέρδη. Αυτές οι νέες εξελίξεις αλλάζουν τη φύση του οργανωμένου εγκλήματος που αυτή τη στιγμή βασίζεται σε μια οργανωμένη δικτυωμένη κοινότητα εγκληματικών ομάδων. Η κατάσταση είναι πολύ πιο ρευστή από ό,τι παλαιότερα. Υπάρχουν ακόμα μεγάλες μαφιοζικού τύπου οργανώσεις, αλλά και νέου τύπου κοινότητες πιο κινητικές εγκληματικών ομάδων. διεθνώς οργανωμένων. Παραδείγματος χάρη οι απομιμήσεις, τα νέα ψυχοτροπικά φάρμακα που λέγονται legal highs και διάφοροι τρόποι κατάχρησης πράξεων από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Αυτά όλα οδήγησαν σε αλλαγές στην εγκληματική αγορά ή στην αγορά του εγκλήματος. Υπήρξε εκμετάλλευση των νέων δυνατοτήτων που δίνει η κρίση για το έγκλημα, ιδιαίτερα η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και καταναλωτριών. Τελεία. Τώρα για μία μικρή ανάλυση των κύριων εγκληματικών τομέων. Τα δρακωτικά είναι ακόμη ο μεγαλύτερος εγκληματικός τομέας και αντιπροσωπεύουν ακόμη το 30% των εγκληματικών δραστηριοτήτων και το λαθρεμπόριο μέσα στην Ένωση Ναρκωτικών συνεχίζει να είναι δυναμικό. Βλέπουμε ότι οι καταναλωτές όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν πολλά είδη ναρκωτικών και όχι ένα. Και γι' αυτό οι ομάδες λαθρεμπορίου έχουν διαφοροποιήσει το εμπόριό τους Τώρα πρόκειται για λαθρεμπόριο πολυναρκωτικών ή πολυλαθρεμπόριο ναρκωτικών. Ε, η ζήτηση ηρωίνης έχει κάπως μειωθεί στην Ένωση, αλλά αυξάνεται η πώληση αφγανικής ηρωίνης μέσω της Ρωσίας. Η... Δεν υπάρχει όμως πια κολομβιανό μονοπόλιο Υπάρχουν μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών σήμερα που συντονίζουν την αγορά. Δεν λειτουργούν ακόμη σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη, αλλά δεν θα αργήσει αυτό. Για την κάναβη, η Ολλανδία παραμένει το κέντρο, εκεί αυξάνεται η ζήτηση, αλλά και αλλού, μέσα και έξω από την Ένωση. Τα συνθετικά ναρκωτικά όμως είναι εκείνα που, όπου σημειώνονται οι περισσότερες και δυναμικότερες εξελίξεις και ιδίως των νέων ψυχοτρόπων φαρημάκων τα οποία μάλιστα καμιά φορά πολλούνται από το ίντερνετ με, γιατί οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται νομικά κενά. Δεν υπάρχει τρόπος ας πούμε να απαγορευθούν, γίνεται να απαγορευθούν, αλλά είναι πιο δύσκολο όταν πολλούνται στο ίντερνετ ενώ παράλληλα νόμιμα πολλούνται με υπό άλλη ετικέτα και καταναλώνονται καμιά φορά από πολίτες εν τη αγνία των ε, τρομερών και θανατηφόρων συνεπειών. Αυτό είναι το καινούργιο κόλπο, αλλαγή του ονόματος. η παράνομη μετανάστευση τώρα οι οικονομικές ανισότητες που συνεχίζονται και αυξάνουν οδηγούν την παράνομη μετανάστευση σε αύξηση προς την Ένωση. Μάλιστα και οι διαφορές μεταξύ των χωρών μελών προς την ενεργεία τους ή τα την κοινωνική περίθαλψη επίσης επηρεάζουν το θέμα. Υπάρχει αυξημένη κατάχρηση των νομίμων οδών με τις οποίες μπαίνουν οι μετανάστες στην Ευρώπη αλλά υπάρχει και εμπορία ανθρωπίνων όντων. Δουλεμπόριο δηλαδή όπου οι παράνομοι μετανάστες υποχρεώνονται να δουλεύουν από εκείνους που τους οργάνωσαν την μετανάστευση, για εκείνους υπάρχει όχι μόνο εργασιακή αλλά και σεξουαλική εκμετάλλευση και η κρίση έχει αυξήσει την ανάγκη για περισσότερα εργατικά χέρια με φτηνότερους μισθούς. τα συστήματα κοινωνικής περίθαλψης γίνονται στόχος των δουλεμπόρων, μερικοί μάλιστα κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ με το δουλεμπόριο αυτό για να εκμεταλλευτούν οι δουλέμποροι τα, την κοινωνική περίθαλψη που δεν παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί. Η μαύρη αγορά, το είπα και πριν, έχει αυξηθεί ιδιαίτερα ως προς τις απάτες και τις απομιμήσεις προϊόντων που έχουν σχέση με τον υγειονομικό τομέα. Πολλοί πέθαναν από την κατανάλωση τέτοιων πλαστών προϊόντων όπως παρελαγμένου εινοπνεύματος στην Τσεχία. Επίσης έχουν χαθεί δισεκατομμύρια από δασμούς που δεν πληρώθηκαν και έτσι στρεβλώθηκε και η ανταγωνιστικότης της, της αγοράς. Αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους εγκληματίες γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση για φτηνά αγαθά. Το εμπόριο απομιμήσεων είναι κάτι που αποφέρει ψηλό κέρδος. Ιδίως αν πρόκειται για, θέμα, για ε, αντικείμενα ή εμπορεύματα πολυτελείας την απάτη των οποίων, την απομίμηση των οποίων ανέχεται περισσότερο και η κοινωνία. Έχουν αυξηθεί λοιπόν τέτοιου είδους προϊόντα απομιμήσεις. Οι οργανωμένες ομάδες επίσης κλέβουν περισσότερο, διενεργούν εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και οι ομάδες αυτές είναι πολύ κινητικές, χρησιμοποιούν, είναι μικρές αλλά κινούνται σε πολλές χώρες και έτσι δυσκολεύεται η δουλειά της αστυνομίας. Και αυτό έχει οικονομική επίπτωση βέβαια και στρέβλωση της αγοράς. Η απάτη και η απομίμηση σας είπα ότι είναι σε αύξηση και αυτό οφείλεται στην κρίση. Τρία στοιχεία κυρίως ελκύουν τους εγκληματίες εδώ. Ο χαμηλός κίνδυνος και η ευκολία με την οποία μπορούν να διαπραχθούν τα αδικήματα αυτά. Υπάρχουν πέντε είδη κυρίως απάτης και στο ίντερνετ και στην κανονική αγορά και φορολογική και δασμολογική απάτη. Οι απάτες αυτές που εμείς ονομάζουμε εκεί με το ακρονίμιο EMTIC αποφέρει πάρα πολύ ψηλά κέρδη. Υπάρχουν και ηλεκτρονικές απάτες για την αποφυγή της πληρωμής του ΦΠΑ. Έτσι χάνονται δισεκατομμύρια από αποφυγή. Οι δασμοί που δεν πληρώνονται συμπεριλαμβάνουν το πετρέλαιο, τον καπνό και το ενόπνευμα. Δισεκατομμύρια λαθε... τσιγάρων έχουν, έχει φανεί ότι πολλούνται παράνομα. Το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος επίσης είναι ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτός από οργανωμένες ομάδες υπάρχουν και επαγγελματικά πλυντήρια βρωμίκου χρήματος η αύξηση του αριθμού των δημοσιονομικών προϊόντων στο ίντερνετ μέσα και έξω από την Ένωση δίνει πρόσθετες ευκαιρίες στους εγκληματίες να ξεπλύνουν το χρήμα των. Το δε κυβερνοέγκλημα επίσης αυξάνεται και αφορά όλες τις χώρες και όλους τους πολίτες. Αφορά ιδιαίτερα δημοσιονομικές απάτες. 8% των χρηστών στο ίντερνετ έχουν ζήσει την εμπειρία κλοπής της ταυτότητός τους. Οι εγκληματίες αυτή τη στιγμή προσφέρουν και ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε άλλους εγκληματίες για τη διευκόλυνση της παρανομίας. Είναι το έγκλημα ως υπηρεσία, ως εξυπηρέτηση. Εν τω μεταξύ και η σεξουαλική κατάχρηση, χρήση παιδών ιδίω αυξάνεται στο ίντερνετ. Γιατί τα παιδιά ευχαρίστως κινούνται στο ίντερνετ και γίνονται εύκολα θύματα. Και στο facebook και twitter φαίνεται αυτό. και εγκλήματα με πιστοτικές κάρτες. 60% των εγκλημάτων πληρωμής οφείλονται στις πιστοτικές κάρτες, ένα δισεκατομμύριο ευρώ περίπου. Και σε, μερικά, σε μερικές χώρες μέλη οι απώλειες ή κλοπές καρτών έχουν αυξηθεί. Νομίζουμε ότι οι εγκληματικές ομάδες συνεχώς θα βρίσκουν καινούργιες ιδέες και τρόπους για να καταχρώνται των online πληρωμών. Επίσης, η αύξηση του αριθμού των αποβλήτων και υψηλή τιμή της απόθεσής τους επίσης ελκύει τους εγκληματίες μπορούν να προσφέρουν φτηνότερες υπηρεσίες απόθεση αποβλήτων, ιδίως στην Δυτική Αφρική και την Ασία. Μερικά συμπεράσματα τώρα. Τα περισσότερα εγκλήματα που εξετάσαμε δεν είναι καινούρια, αλλά αυτό που εντυπωσιάζει είναι η εξέλιξη των εγκληματικών δραστηριοτήτων και η βιωσιμότητα των ίδιων των εγκληματικών ομάδων. Τουλάχιστον 3.000 από αυτές παραμένουν και αποτελούν σημαντική απειλή για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες στην Ένωση. Είναι πολύ καινοτόμες και ευέλικτες. Εκμεταλλεύονται όλες τις ευκαιρίες που μπορεί να τους δοθούν ιδίως, ιδίως λόγω της κρίσης. Εκτός από αυτήν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες στην κοινότητα που διευκολύνουν το έγκλημα. Οι νέες τεχνολογίες, το ίντερνετ και οι διάφορα κενά στην νομοθεσία. Γι' αυτό φέτος αφιερώσαμε ολόκληρο κεφάλαιο στην ανάλυση αυτών των νέων δυνατοτήτων για το έγκλημα και σημαντικό είναι του χρόνου όταν θα το ξαναδούμε να εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε να μειώσουμε τις ευκαιρίες αυτές, τις αυξημένες ευκαιρίες που έχουν οι εγκληματίες από τη σύγχρονη κοινωνία. Ο συνάδελφός μου τώρα, πρόεδρος της Κόζη, θα σας μιλήσει σε λίγο για τη σημασία της έκθεσης αυτής μέσα στα πλαίσια της νομοθέτησης ή του κύκλου νομοθεσίας της ε, Ένωσης. Εγώ θα τελειώσω με ορισμένα, ορισμένες συστάσεις για τους νομοθέτες. Πρώτον, νομίζω ότι η μελέτη μας δείχνει ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι μεγάλη απειλή για την κοινωνία και γι' αυτό θα πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητες της Ένωσης. Έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ζωή των επιχειρήσεων και των πολιτών και διαφοροποιείται συνεχώς. Το τελευταίο ευρωμαρόμετρο έδειχνε ότι 25% των πολιτών τουλάχιστον ανησυχούν από την αύξηση του οργανωμένου εγκλήματος και ιδιαίτερα για την εμφάνιση του κυβερνοεγκλήματος. Φυσικά ξέρουμε ότι τα κονδύλια που αφιερώνονται στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος από τον νοσιακό προβληματισμό είναι πολύ χαμηλά. Και αναρωτιέται κανείς λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στις ευχές των πολιτών μας με τόσο λίγα λεφτά. Επίσης για τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε μια ενοποιημένη προσέγγιση ως ανταπόκριση στο οργανωμένο έγκλημα. Έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις εδώ στην οικονομία. Αυξάνεται η μαύρη αγορά, αυξάνονται οι ζημίες, και οι απάτες. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη και για την επιτυχή καταπολέμηση του οργανωμένου εγκουλήματος. Αν θέλουμε η οικονομία στην Ευρώπη να αναπτυχθεί. Πώς, θα πώς να διευθετηθεί το ίντερνετ είναι θέμα πάρα πολύ ακανθόδες εδώ και καιρό. Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Πάντως από πλευράς επιβολής του νόμου ξέρουμε ότι το ανοιχτός χαρακτήρας του ίντερνετ είναι τεράστια ευκαιρία για τους εγκληματίες και οι επιπτώσεις του εγκλήματος ψυχολογικά ή σε άλλους τομείς όπως για τη σεξουαλική εκμετάλλευση και αυτές αυξάνονται παραπάνω από τις δυνατότητες, νομοθετικές μας δυνατότητες. Ας πούμε η σύμβαση της Βουδαπέστης είχε υπογραφεί ήδη πριν από 10 χρόνια και από τότε οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Τώρα η σημασία της διεθνούς συνεργασίας βλέπουμε ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες και συμπεριφορές κινούνται από το εθνικό στο διεθνές επίπεδο. ομάδες που δρούσαν σε ένα μόνο κράτος δεν υπάρχουν σχεδόν πια. Στη μελέτη μας βρήκαμε ομάδες που έχουν περίπου, αποτελούνται από πάνω από 60 εθνικότητες και δρούν σε 35 χώρες. Αυτό είναι ο νέος τύπος του οργανωμένου κλίματος. Πολύ διεθνιστικού χαρακτήρος. Και άρα διεθνής πρέπει να είναι και η ανταπόκριση, η αντιμετώπιση. Πολύ περισσότερη συνεργασία λοιπόν χρειάζεται στην Ένωση για να το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, σας κατευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αλλά πριν να, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα δώσω το λόγο στον Μαρτίν Πάουερ, ο οποίος είναι επικεφαλής, είναι πρόεδρος της Κόσεφ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να σας πω καταρχήν ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας να απευθυνθώ σε σας σήμερα εκ μέρους της ομάδας Κόζη. Είμαι επικεφαλής του Τμήματος Ασφαλείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ε, στο Δουβλίνο και είμαι και πρόεδρος της ε, ΚΟΖΙ στα πλαίσια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Ε, να παρουσιάσω κάποιο από το background της ΚΟΖΙ, κάποιο από το έργο της και το ρόλο της σε σχέση με τον κύκλο πολιτικής. Όπως είπατε και στην αρχή, ξεκινάμε τώρα ένα νέο κύκλο πολιτική. επομένω είναι σκόπιμο ε, να σα τα παρουσιάσω αυτά εγώ σήμερα. Το 2013 είναι η τέταρτη χρονιά εργασία τη ΚΟΖΗ, συστήθηκε από απόφαση του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου του 2010 μετά από τη δημιουργία μιας ομάδας ΚΟΖΗ δυναμή του άρθρου 71 της Συνθήκη τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια επιτροπή υψηλού επίπεδου, πρόκειται για μια, μια ομάδα εργασία του Συμβουλίου, αλλά ο στόχο είναι να προωθήσει και να ενδυναμώσει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών τη Ευρωπαϊκή Πένωση στον τομέα τη εσωτερική ασφάλεια. Αυτή είναι μια ευρεία έννοια η έννοια τη εσωτερική ασφάλεια εδώ δεν διεξάγει δικές της επιχειρήσεις, ούτε έχει νομοθετική λειτουργία. Επικεντρώνεται αποκλειστικά στο να διασφαλίσει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών και των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση του εγκλήματος οργανωμένου και μη. Υπάρχει και το Συμβούλιο ΔΕΗ που υποστηρίζει ε, την ομάδα τη της Βρυξέλλες. Επίσης υπάρχει και μια σειρά υπηρεσιών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στην κόζη όπως η Europol, η Frontex, η Σεπόλ και η Eurojust μεταξύ άλλων συνδέονται πολύ στενά με τις δραστηριότητες της ΚΟΖΗ και συμμετέχουν σε θέματα της ημερησίας διάταξης που τους αφορούν. Ενίοτε, οι εκπρόσωποι από άλλους οργανισμούς όπως η ΟΛΑΦ, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο όπως και ε, ο Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων επίση συμμετέχουν. Συνήθω έχουμε δύο-τρει ε, συνεδριάσεις, ένα προεδρία, δηλαδή ετησίω περίπου πέντε συνεδριάσεις και συζητάμε μαζί με την ε, Επιτροπή Πολιτική σε κοινά θέματα. Έχουμε διαδραματίσει τρει, έχουμε συγγνώμη, προγραμματίσει τρει συνεδρίας τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Η μία χώρα, οι δύο θα λάβουν χώρα στο μέλλον, αλλά σε σχέση με τις απειλέ ε, στο Μαλί και στην Αλγερία και ε, τα γεγονότα στην Αλγερία τον Ιανουάριο με τις απαγωγές η Κόζη συνεδρίασε έκτακτα στις 28 Φεβρουαρίου για να συζητήσει τις απειλέ από τη Βόρεια Αφρική προκειμένου να προετοιμάσει συμπεράσματα του Συμβουλίου για το Συμβούλιο ΔΕΗ που επίση έλαβε χώρα τον ε, Φεβρουάριο, μάλλον αρχές Μαρτίου. Ποιο ε, είναι τώρα το πεδίο δράση τη ΚΟΖΟ, ποιο είναι ο στόχο, είναι να διασφαλίσει την αποτελεσματική συνεργασία και το συντονισμό στον τομέα τη εσωτερική ασφάλεια, αστυνομία, τελωνία, συνοροφύλακε και δικαστικέ αρχέ, που όλοι δραματίζουν ένα ρόλο σε αυτό το τομέα επίση. Αξιολόγηση τη γενική κατεύθυνση και αποτελεσματικότητα τη επιχειρησιακή συνεργασία και να βοηθήσει το Συμβούλιο σε σχέση με τη ρήτρα αλληλεγγύης δυνάμεις του άρθρου 222 της Συνθήκης. Οι βουλευτές θα γνωρίζουν ότι πρόσφατα η δεύτερη έκθεση της ομάδας Κόζη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια διαβιβάστηκε κατόπιν έγκριση του Συμβουλίου. Η έκθεση αυτή κάλυπτε τις δραστηριότητες της ΚΟΖΗ κατά το προηγούμενο τρίου των Προεδριών Πολωνία, Δανία, Κύπρος και καλύπτει και την περίοδο από τον ε, Ιούλιο του 2011 μέχρι τα τέλη του 2012. Μέχρι τώρα εστιάστηκε η ΚΟΖΗ κυρίως στο κύκλο πολιτικής ε, και αυτό αφορά διάφορους τομείς, να καθοριστεί η μεθοδολογία για την ανάπτυξη του κύκλου πολιτικής, να δοκιμαστεί ο κύκλος πολιτικής, να εφαρμοστούν τα οποιαδήποτε διδάγματα και τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της ανάπτυξης ενός νέου κύκλου πολιτικής. Υπάρχουν κάποια κύρια βήματα σε αυτό το κύκλο πολιτικής. Καταρχήν η αξιολόγηση των απειλών. Αυτό κάνει η Europol και αυτό μόλις ακούσαμε από το διευθυντή της Europol. Κατόπιν η χάραξη της πολιτικής. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο που εμπλέκεται η κόζη στην ε, εκπόνηση συμπερασμάτων και κατόπιν ε, έχουμε το στάδιο της εφαρμογής που σε μεγάλο βαθμό αφορά τα κράτη-μέλη, ε, να το εφαρμόσουν σε συνεργασία με τη Europol και κατόπιν να έχουμε την αξιολόγηση από την οποία θα προκύψει ο επόμενος κύκλος πολιτικής και ίσως να έχουμε καλύτερη εστίαση σε κάποιους τομείς. Βάσει της ε, μελέτης ε, της αξιολόγησης απειλής ε, για το οργανωμένο έγκλημα του 2011 περιλαμβάνοντας την κύκλο πολιτικής, το έγκλημα στα Δυτικά Βαλκάρια και το οργανωμένο έγκλημα γενικά εμπορία ανθρώπων κτλ σε περιφερειακή βάση επικεντρωνόμαστε σε περιοχές όπως η Δυτική Αφρική και τα Δυτικά Βαλκάνια, ε, όπου είχαμε εγκλήματα που έφυγαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης επικεντρωθήκαμε σε κάποια συγκεκριμένα εγκληματικά φαινόμενα όπως η λαθρομετανάστευση, η εμπορία ανθρώπων, τα ναρκωτικά, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Αυτά που ακούσαμε να μας αναφέρει ο Διευθυντής της Europol, αλλά εξακολουθούν φυσικά ναι, υπάρχουν και σήμερα σημαντικοί παράγοντες και υπάρχουν και οριζόντιες πτυχές, ε, όπως ε, παραδείγματο χάρη να δούμε τι διευκολύνει το έγκλημα σε διάφορους τομείς. Ε, τα κράτη-μέλη θα συμμετείχαν στις συνεδρία της ΚΟΖΗ και θα λειτουργούσαν ως κινητήριες δυνάμεις και θα συμμετείχαν τα κράτη-μέλη αλλά και οι οργανισμοί όμως ε, θεωρήθηκε ότι ήταν καλό να διοριστούν κάποιοι άνθρωποι που θα καθοδηγούν τη δουλειά σε αυτούς τους τομείς και κατόπιν οι προτεραιότητες μεταφράστηκαν σε στρατηγικούς στόχους και σε επιχειρησιακά σχέδια δράσης για να εντοπιστούν συγκεκριμένες δράσεις που έπρεπε να αναλυφθούν για να υπάρξουν και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στην επόμενη συνεδρίαση της ΚΟΖΗ, όπως είπε η της Europol, η ΚΟΖΗ θα κάνει ένα παρόμοιο εγχείρημα. Δηλαδή θα προσδιορίσει τις κύριες απειλές και θα εκπονήσει συμπεράσματα του Συμβουλίου. Η μεθοδολογία ΣΟΚΤΑ αναπτύχθηκε μέσω της ΚΟΖΗ το 2012 και είχε σχεδιαστεί για να παρουσιάσει τις ε, ε που διέπουν την ΟΚΤΑ. Ε, παρήχαμε τη μεθοδολογία για την εκπόνηση της έκθεσης και παρουσιάσαμε τι αναμενόταν να προκύψει από τη ΣΟΚΤΑ και πώς θα έπρεπε να μοιάσουν τα συμπεράσματα στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Ένα μέρος αυτού είναι να διασφαλίστη ότι οι προτεραιότητες που θα καθοριστούν είναι αυτές που τα κράτη-μέλη, οι οργανισμοί και το Συμβούλιο πιστεύουν ότι είναι αυτές που απαιτούν περισσότερη προσοχή. Σε ό,τι αφορά στην παρακολούθηση της διαδικασίας, υπό την Προεδρία της Δανίας είχαμε μια αναθεώρηση της διαδικασίας του πρώτερου κύκλου πολιτικής. Επικεντρώθηκε κυρίως στα όσα έκανε η Κόζη γενικά η παρακολούθηση προόδου έγινε βάσει των σχεδίων δράσης. Υπήρχε λοιπόν συνεισφορά από όσου έδιναν όθηση στις προτεραιότητες στους εθνικούς συντονιστές και τη Europol. Επίσης, είχαμε και ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που αξιολογούσε το κύκλο πολιτικής για να παρέχει ενημέρωση για την ανάπτυξη του επόμενου κύκλου πολιτικής. Τα κύρια πορίσματα ήταν εξακολουθήσε να υπάρχει γενική εντύπωση ότι ο κύκλο πολιτική είχε προστιθέμενη αξία. Υπήρξε σαφή μεθοδολογία που είχε καθοριστεί στην εφαρμογή και την αξιολόγηση των προτεραιών για την αξιολόγηση των σοβαρών απειλών Επίση, ε, υπήρχε εμπειρία στις συνεργασία για την επίτευξη των προτεραιοτήτων μεταξύ διάφορων πρωταγωνιστών ε, και είδαμε και ξεκάθαρο ρόλο της Europol. Υπήρξαν τομεί όπου προσδιορίστηκαν, εντοπίστηκαν ε, κάποιε βελτιώσει για να μπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα. Ένα τομέα ήταν να προσπαθήσουν να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν περισσότερο, γιατί αν συμμετέχουν τα κράτη-μέλη τότε τα αποτελέσματα σίγουρα θα βελτιωθούν, γιατί πρέπει να δούμε τι πιστεύει το κράτο μέλος ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια του εγκλήματος. Φυσικά συμμετέχουν τα κράτη-μέλη και οι εκπρόσωποι τους διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο προς τη θέσπιση των στόχων. Πρέπει να υπάρξει και πρόθεση της ε, ευαισθησίας σε σχέση με τον κύκλο πολιτικής, ε, δηλαδή στα κράτη-μέλη πρέπει να γίνει πιο γνωστός ο κύκλος πολιτικής, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο οι στην καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος και η ΣΕΠΟΛ διαδραματίζει ένα ρόλο στο να αναπτύσσει πακέτα για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος. Επίσης, θεωρήθηκε ότι υπήρχε ανάγκη για πιο συγκεκριμένη διατύπωση των στρατηγικών στόχων και αυτό για να διασφαλίσει ότι οι δράσει, τα ετήσια σχέδια δράση ήταν επαρκώ επιχειρησιακέ. Σε μεγάλο βαθμό αυτό θέλουμε να κάνουμε, ότι δηλαδή πραγματικά λειτουργούν αυτά τα σχέδια, γιατί μόνο έτσι η κόζη μπορεί να αξιολογήσει αποτελεσματικά. Επίση, θεωρήθηκε ότι η ΕΕ έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρηματοδότηση, αλλά και σε άλλου τομεί. και αυτό ήταν ζωτικό για την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων δράση. Και όπως αναφέραμε ήδη, ξεκινά με ένα νεοκυκλοπολιτικής, η ΣΟΚΤΑ μόλις δημοσιεύτηκε και ο ρόλος της ΚΟΖΗ θέλει να την εθετήσει να θέσει τις προτεραιότητες, που είναι ο κύριος στόχος της επόμενης συνεδρίας τον Απρίλιο, και από εκεί και πέρα να καταλήξουμε σε συμπεράσματα του Συμβουλίου για το Συμβούλιο του Ιουνίου. Επομένως, ε, φυσικά ερχόμαστε σήμερα εδώ σε μια πολύ κατάλληλη χρονική στιγμή να σας τα αναφέρουμε όλα αυτά. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στη διαδικασία να ε, περιμένουμε τις απαντήσεις των κρατών μελών για τη ΣΟΚΤΑ πριν να καθορίσουμε την ατζέντα της ΚΟΖΗ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να τοποθετηθώ επί της ΣΟΚΤΑ αλλά η ΚΟΖΗ πρέπει να προσδιορίσει τους διάφορους πρωταγωνιστές όπως και τις διάφορες προτεραιότητες και ε, φυσικά θα καθοριστούν ποιοι θα οθήσουν αυτές τις προτεραιότητες. Θα καθοριστούν πολυετή στρατηγικά σχέδια για κάθε προτεραιότητα και κατόπιν θα έχουμε τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης. Επομένως, η ΚΟΖΗ θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να λαμβάνει εκθέσεις για την εφαρμογή των σχεδίων δράσης. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τομείς και είδη εργασίας όπου εμπλέκεται η κόζη, όπως ε, το χάρη στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τα Ναρκωτικά. Εκεί έχουμε μία σειρά από ομάδες ε, project για να εφαρμοστούν οι δράσεις για την καταπολέμηση του εμπορίου ειρήνης κοκαίνης, οργανωμένου εγκλήματος κτλ. Παρακολουθεί δραστηριότητες και αποφασίζει Ποιε από τι δραστηριότητες είναι καλύτερο να συνεχιστούν για την κοκαίνη και την ηρωίνη παραδείγματο χάρη στι διάφορες επιχειρήσεις και στα σχέδια δράση και στα έσοδα και για τα έσοδα από το οργανωμένο έγκλημα. Ε, ενισχύουμε την προστασία των ε, εξωτερικών συνόρων για καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Πώς? Με την σύσταση 5 μέτρων. Εμείς θεωρήσαμε ότι μπορούσαν να συνεχιστούν κάποιες δράσεις για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και επίσης η ΚΟΣ ζήτησε να υπάρξουν σχέδια δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των μεταναστευτικών πιέσεων για τη Δυτική Αφρική. συντονίσαμε δράσεις για την καταπολέμηση του κλίματος στη Δυτική Αφρική, το παρακολουθήσαμε αυτά και δώσαμε καθοδήγηση σε σχέση με τα μέτρα που είχαν προσδιοριστεί για την καταπολέμηση του εγκλήματος που προέρχεται από αυτή την περιοχή. Επίσης, υπήρξε συνεισφορά από Europol και Σεπόλ για την ανταλλαγή απόψεων για τι επιχειρησιακέ απαιτήσει για το μέλλον Europol και ΣΕΠΟΛ. Σε σχέση με το συντονισμό, ο ρόλος της ΚΟΖΗ είναι να διασφαλίσει και να διευκολύνει τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών ΔΕΗ, των οργανισμών ΔΕΗ. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την ΚΟΖΗ. Και υπάρχει μια ετήσια συνεδρίαση των επικεφαλής αυτών των υπηρεσιών και αναφέρουν στην ΚΟΖΗ Πώ έχουν συντονίσει τι δικέ του απαντήσει στα διαφορά κλιματικά φαινόμενα. Υπάρχει επίση συνεργασία με την, εξωτερική, με την πτυχή εξωτερικής ασφάλειας υπάρχουν συνεδριάσεις μεταξύ της ΚΟΖΙ και την Επιτροπή Πολιτικής Ασφάλειας για να ενδυναμωθεί η συνεργασία και ο συντονισμός ε, σε όλα τα θέματα της ασφαλείας και στις εξωτερικές πτυχές. Και ανέφερα και το τι ανέκυψε στο Μάλι, στη Βόρεια Αφρική και στην Αλγερία ε, νωρίτερα φέτος. Συζητήθηκε αυτό το θέμα σε μια κοινή συνεδρίαση ΚΟΖΗ και Επιτροπής Πολιτικής Ασφάλειας. Επίσης, η αξιολογεί την έκθεση της Κομισιόν για την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Το δεύτερο έγγραφο θα παρουσιαστεί τον Απρίλιο στις συνεδρίες της ΚΟΖΗ. Αξιολογήσαμε τον προηγούμενο κύκλο, προετοιμάζοντας ε, το νέο κύκλο. Επίσης, ε, η ΚΟΖΗ εξετάζει μια σειρά άλλων εκθέσεων, όπως ε, την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την παράνομη εμπειρία κτλ. Η Κόζη ουσιαστικά έχει μάθει πολλά, έχει πολλά διδάγματα από τον πρώτο κύκλο πολιτικής που καλύπτει την προηγούμενη περίοδο και έχει αναπτύξει μία μεθοδολογία για να αναπτύξει τη σημερινή σόκτα και τώρα θα προβεί σε εφαρμογή, θα την παρακολουθήσει και κατόπιν θα προκύψει ένας νέος κύκλος πολιτικής. Δεν έχω να πω πολλά παραπάνω. Ελπίζω να σας έδωσα κάποια ιδέα για το πώς λειτουργεί η κόζη. Να τονίσω όμως ότι η Προεδρία δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο τριμερή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλους αυτούς τους τομείς. Και φυσικά ενδιαφέρομαι πάρα πολύ να ακούσω και τις απόψεις σας για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε τον κατάλογο μιλητών, κυρία Ματιέ, Άλμπρεχτ, ο κύριος Παπα-Νικολάου και δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλο να πάρει το λόγο. Κύριε Ματιέ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον κύριο Βέινράιτ για την καταπληκτική μελέτη που μας παρουσίασε Αλλά δεν χρειάζεται απεσιοδοξία, τόση απεσιοδοξία, γιατί αν ισχύουν αυτά αυτά όπως τα είπατε πρέπει να πάμε όλοι να πέσουμε από το παράθυρο. Ξέρετε ότι είμαι μέλος της επιρικής Επιτροπής Καταπολέμησης του Εγκλήματος. Σας έχουμε συναντήσει εκεί και άλλες φορές και τους συνεργάτες σας, αλλά οι ακροάσεις μας και οι μελέτη δείχνουν ότι τα πράγματα είναι αρκετά μαύρα και μέσα στην Ένωση, όχι μόνο εκτός. Όλα αυτά δεν είναι και πολύ καλά για να μας υψώσουν το ηθικό. Η μαύρη αγορά, κοιτάξτε, όλοι βλέπουμε λίγο πολύ πώς λειτουργεί η μαύρη αγορά, δεν μας εκπλήσει ότι αυξήθηκε, αλλά Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο είναι αυτά που είπατε για την ε, παιδεραστία που λέτε ότι χειροτερεύει και ότι εμείς οι νομοθέτες έχουμε αποτύχει καθώς και οι αστυνομικές και οι άλλες διοκτικές αρχές και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε όντως για τα παιδιά βέβαια, αλλά και για τους νέους γενικότερα οι οποίοι είναι τοξικομανιστή, κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτά που λέει η μελέτη σας είναι πολύ ανησυχητικά. Καθώς και το δουλεμπόριο και αυτό πολύ ανησυχητικό. Μας μιλήσατε και για περιβαλλοντολογική εγκληματικότητα. Κάποιος συνεργάτης σας είχε έρθει στην Επιτροπή καταπολέμησης που μας είπε και εκείνος πολύ ανησυχητικά πράγματα για απομιμήσεις ε, ζυζανιοκτώνων, παρασιτοκτώνων που χρησιμοποιούν οι γεωργοί με τρομερές συνέπειες στην υγεία και άλλα προϊόντα γιατί φαίνεται ότι οι εγκληματικές ομάδες ε, προσαρμόζονται πάρα πολύ γρήγορα στην εξέλιξη της αγοράς και μάλιστα καλύτερα από τους νομοθέτες και του, τις διοκτικές αρχές και τους δικαστάς. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, έχετε καμιά λύση ή ο κύριος Πάουερ της Κόζη. Τρομακτικά όλα αυτά. Και τέλος, μας μιλήσατε και για ελαθρεμπόριο όπλων. Ξέρουμε τα όπλα τύπου Καλάσνικοφ που προέρχονται από τα Βαλκάνια και που τα βρίσκουμε μέχρι και στη Γαλλία για... και χρησιμοποιούνται κυρίως από τη μαφία. Για αυτού του τύπου τα όπλα έχετε αριθμούς. Γιατί μας λέτε ότι υπάρχει λαθρεμπόριο όπλων και νόμιμο. Ε, τότε πώς είναι λαθρεμπόριο, τέλος πάντων, τα οποία Διακινούνται όμως κρυφίως, νόμιμο αλλά κρυφά. Έχετε αριθμούς και για αυτά. Τι όπλα είναι αυτά. Τι όπλα είναι. Μερικά είναι λέει αστυνομικά όπλα. Εξουδετερωμένα. Τα οποία μετά πολλούνται, κυκλοφορούν. Μήπως έχετε καμιά λεπτομέρεια για αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία μου. Επόμενος ομιλητής, Άλμπρεχτ, μπείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον, κύριο Ρέινράιτ και τον κύριο Πάουρ για την ε, παρουσίαση που μας κάναν. Πολύ συνοπτική, σας ευχαριστούμε. Δύο ερωτήσει να κάνω σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία συζητάμε γιατί θα με βοηθούσε πάρα πολύ. Και θα μας βοηθούσε και στη δουλειά μας. Να έχουμε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, ενημερωμένα για τα ποσοστά εγκληματικότητας και σε ό,τι αφορά το ύψος ε, του ξεπλήματος χρήματος, το, της απάτης. Ξέρω ότι δεν χρειάζεται να μπείτε σε λεπτομέρειες, απλά θα ήθελα να έχουμε παραπάνω λεπτομέρειες εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και στην Επιτροπή ΚΡΙ, ασφαλώς. Το δεύτερο θέμα, μία ερώτηση για τώρα. Σε ποιους ορισμούς βασιζόμαστε όταν μιλάμε για τις κατηγορίες αυτές. Γιατί αυτό πολλές φορές το συζητάμε για το έγκλημα αλλά και για άλλους τομείς και σε κάποια φάση θα πρέπει να έχουμε κοινού ορισμούς για να ξέρουμε τι ακριβώς συζητάμε. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω, αν έχετε κάτι να μας πείτε, προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε τους ορισμούς αυτούς, καθώς αντιμετωπίζουμε καινούριου ε, κανόνες και την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου. Είναι πιο σημαντικό παραποτέ να υπάρχουν σαφείς ορισμοί. Και σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για το ποινικό δικαίωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα έχουμε τον Γιάννη Μούλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτά που μας παρουσίασε ο κύριος Wainwright ήταν πάρα πολύ απεσιόδοξα και μαύρα για το μέλλον μας και όσο πιο πολλά στοιχεία άκουγα τόσο πιο απεσιόδοξος γινόμουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει ελπίδα, αλλά όπως και να έχει η κατάσταση κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Πρώτη ερώτηση λοιπόν, η Europol έχει στην παρούσα φάση αρκετές ε, αρμοδιότητες ε, προκειμένου να μπορέσει να δράσει ή θα ήθελε παραπάνω αρμοδιότητε, γιατί θα μπορούσαμε ενδεχομένω στο Κοινοβούλιο να βοηθήσουμε. Είναι ικανοποιητική η τρέχουσα κατάσταση ή πρέπει να προσθεθούν και αρμοδιότητε. Και επίση πολύ συχνά αναφερθήκατε στο έγκλημα στο διαδίκτυο και ότι κατίσταται, καθίσταται όλο και περισσότερο μέσο για τέτοια εγκλήματα ως χρήσης του ίντερνετ. Αναρωτιέμαι τι μπορούμε να βοηθησουμε ειναι ικανοποιητικη η τρεχουσα κατασταση η πρεπει να προσθεθουν και αρμοδιοτητε και επιση πολυ συχνα αναφερθηκατε στο εγκλημα στο διαδικτυο και οτι κατηστατε καθισταται ολο και περισσοτερο μεσο για τετοια εγκληματα ως χρησης του ιντερνετ αναρωτιεμαι τι μπορουμε να κανουμε αν τέτοια πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο και εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε κάτι να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε Γιάν, λέει ο Πρόεδρος και πρωτού δώσω το λόγο στους δύο πανελίστες εξ αριστερών. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για το οργανωμένο έγκλημα ε, αξιωματούχοι της Φιλανδικής Κυβέρνησης ε, μου ανέφεραν ότι διακρίνονται καινούργια ε, και καινούργιε μορφέ και σχήματα εγκλήματος. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν προς τα ποια κατεύθυνση κινούμαστε και τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσει αυτές. Δεν είχα πρόθεση καμία να σας καταθλίψω σήμερα και να δείξω απεσιόδοξία αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ιδιότερα σε θέματα μεθοδολογίας ε, φροντίζουμε να είμαστε αντικειμενικοί και εξαρτώμαστε από τα στοιχεία που μας ε, χορηγούν τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται. Χαιρόμαστε που είναι επαγγελματικό ο τρόπος ε, εργασίας μας. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν που διαμορφώνεται για τα ερωτήματα συγκεκριμένα. Προς την κυρία Ματιό, καταρχάς, να απαντήσω το εξής. Θεωρώ επειδή μιλήσατε για την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο ίντερνετ, ε, οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουμε για την καταπολέμηση του εγκλήματος στο διαδίκτυο, όπου για παράδειγμα οι εγκληματίες μπορούν να καταχρούνται ε, στις ταυτικά στοιχεία του διαδικτύου, όπως η αρχή της ανωνυμίας. Είναι αμέσως αμέσως πάρα πολύ δύσκολο για την αστυνομία να βρει τον εγκληματία. Το γεγονός ότι έχουμε τέτοια τεχνολογικά πλεονεκτήματα που έχουμε πολλά χαρακτηριστικά ασφαλείας online προκειμένου να κρύψει κανείς ε, την ταυτότητά του και τη δραστηριότητά του. Αναδύονται για να μείνω στην απασιόδοξη εικόνα την ανάδεση του Darknet online ένα τμήμα του ίντερνετ το οποίο κρύβεται πίσω από πολλά επίπεδα ε, κρυπτογράφησης και όπου μπορεί κανείς να αποθηκεύσει και να ανταλλάξει τέτοιο υλικό. Απεριόριστες ουσιαστικά δυνατότητες αποθήκευσης με όλο και πιο πολλά τεχνολογικά πλεονεκτήματα κάθε χρόνο και σε ό,τι αφορά την παιδεραστία. Α υποθέσουμε ότι ένας αστυνόμο καταλήγει σε μια διεύθυνση και βλέπει κάποιες φωτογραφίες, βίντεο ενδεχομένω σε κάποιες ε, από τι επιχειρήσει μας βλέπουμε ότι οι ύποπτοι έχουν κατεβάσει megabytes, 44.000 ε, ώρες ε, σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών γιατί όλα αυτά διατίθενται στο διαδίκτυο και έχει γίνει πλέον καθημερινότητα η ανταλλαγή τους και η δυνατότητα να δημιουργηθούν δίκτυα παγκοσμίω τέτοιων εγκληματιών. Και τίφονται και θέματα λοιπόν δικαιοδοσία. Πού ξεκινά, πού σταματάει το ίντερνετ για παράδειγμα. Ένα καλό παράδειγμα λοιπόν όπου οι παραδοσιακοί μέθοδοι ποινική δίωξη έχουν καταστεί ανήμπορες ένα συνοριοφύλακα ο οποίο σταματά για παράδειγμα τον λαθρέμπορο ναρκωτικών δεν μπορεί να το κάνει αυτό online γιατί το σύνορο στην περίπτωση αυτή είναι εικονικό. Και για να συνεχίσουμε ε, επ' αυτού, κύριε Άλμπρεχτ, με ρωτήσατε για τις διαστάσεις του προβλήματος. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι αυτό ε, είναι κάτι το οποίο δυστυχώ που δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Δεν υπάρχει αρκετή έρευνα στην ακαδημαϊκή κοινότητα για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή διάσταση του προβλήματος. Έχουμε κάποιες εκτιμήσεις, ξέρουμε ότι από τις πληρωμές των πιστοτικών καρτών έχουμε 1,5 δισεκατομμυρίων ανά έτος. Ξέρουμε ότι απώλειες λόγω ΦΠΑ είναι 100 δισεκατομμύρια ένα έτος, σύμφωνα με τις εκθέσεις της ε, Κομισιόν και θεωρούμε ότι αυτό εν μέρη οφείλεται σε εγκληματικές ε, στο οργανωμένο έγκλημα. Δεν ξέρουμε τι ποσοστό όμως ακριβώς ε, μιλάμε. Στο κυβέρνο έγκλημα δεν έχουμε καλά ποσοστά, καλά αριθμητικά στοιχεία. Μας δίνουν και οι εταιρείε και ο κλάδος κάποια στοιχεία, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αξιόπιστα αλλά ακόμα και κάποια από τα στοιχεία που διαθέτουμε μας καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι μικρό και ότι αυξάνεται μάλιστα σε ό,τι αφορά τους ορισμούς. Συμφωνώ με τον κύριο Άλμπρεχτ ότι ίσως θα χρειαστεί ένα χτένισμα της μεθοδολογίας μας. Θα θέλαμε τα κράτη-μέλη να μας δώσουν την ερμηνεία του οργανωμένου εγκλήματος. Άρα θεωρούμε ότι μοιραία θα υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές σε ό,τι αφορά την ερμηνεία το οποίο ενδεχομένω να περιορίσει την αξιοπιστία των πορισμάτων μας, αλλά δεν αναμένω μεγάλες διαφορές. Ε, θεωρώ ότι λίγο πολύ, για παράδειγμα, το λατρεμπόριο κοκαίνης ε, έχει τον ίδιο ορισμό σε όλα τα κράτη-μέλη. Για το οργανωμένο έγκλημα ενδεχομένω να υπάρχουν μεγαλύτερες διαφορές. Κύριε Μίλτερ, μας ρωτήσατε για το κατά πόσο το διαδίκτυο και τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτό. Από τη φύση του το πρόβλημα αυτό είναι παγκόσμιο. Είναι περιορισμένες οι αντιδράσεις μας, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ας ε, διασφαλίσουμε ότι υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ προστασίας, ελευθερία ε, του διαδικτύου το οποίο αποτελεί προφανώς ε, ένα, μια αρχή, μια αξία την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε και εγώ ως αστυνομικό ακόμα, αλλά να μην χαθούμε στο διαδικτύο, να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα προκαλείται όλο και μεγαλύτερη ζημιά στις κυβερνητικέ υπηρεσίε στους πολίτες. Τι σημαίνει αυτό, για παράδειγμα, να διασφαλίσουμε ότι η αστυνομία έχει πρόσβαση στις σωστέ πληροφορίε, στη σωστή στιγμή από του παρόχου και θα ήθελα σε κάποιες περιπτώσεις η διεθνής κοινότητα και τα συμφέροντά της να συζητιόνται καλύτερα κατά την ε, κατάρτιση νέας νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την, την ε, οδηγία για την ε, διατήρηση των δεδομένων, την προστασία των δεδομένων, την τεχνολογία του διαδικτύου και του καθεξής. Ο κ. Μίλτερ επίσης ρώτησε αν έχουμε επαρκείς πόρους και αρμοδιότητες στην Europol δεν είναι θέμα αρμοδιότητα. Σωστά κάνουν οι αρμοδιότητε και είναι στα χέρια των εθνικών αρχών. Θεωρώ ότι η Europol θα πρέπει να έχει ανεξάρτητε αρμοδιότητε για την δίωξη των εγκληματιών. Θα πρέπει να υπάρχει διεθνή αντίδραση του προβλήμα, στα, στο πρόβλημα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν λοιπόν αυτό που καλούνται να κάνουν. Δεν είναι θέμα αρμοδιότητα, μπορεί να είναι θέμα όμω πόρων. Και μια και μιλάμε για τα προβλήματα στο διαδικτύο, δεν μπορώ παρά να υποφεληθώ από την ευκαιρία και να σας πω ότι πέρσι αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια, ένα τμήμα για την καταπολέμηση του εγκλήματος στο ίντερνετ χωρίς να του ε, χορηγήσει κονδύλια. Άρα νομίζω ότι αυτό απαντάει το ερώτημά σας. Μας ρωτήσατε για τα νέα, τις νέες μορφές εγκλήματος. Βλέπουμε νέες μορφές εγκλήματος online στο διαδίκτυο. Αυτές που σας περιέγραψα μας ε, ανησυχούν και λίγο, να σας πούμε την αλήθεια, τα εγκλήματα κάτω του περιβάλλοντος, τράφικινγκ από βλήτων. σε ό,τι αφορά τις αγορές ενέργειας ε, και αυτές αποτελούν ένα βασικό τομέα που μας ανησυχεί. Και τέλος, κυρία Ματιέν, μας είπατε για το τράφικινγκ στο διαδίκτυο. Δεν έχω πολλές πληροφορίες, πολύ φοβάμαι ίσως κατεδίαν ε, να σας διαβάσουν τις πληροφορίες αυτές, αν το επιθυμείτε. Ο κύριος. Κύριε Πάουρ, θέλετε να συνεχίσετε. Να κάνω δύο σχόλια, αν μου επιτρέπετε. ο επικεφαλής της Γρούπας αναφέρε κάποια τομείς προτεραιότητες και μία σειρά φαινομένων όπως η απάτη, το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος κτλ. Ανέφερε την ιδέα της ασφάλειας για την ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα από τα θέματα της Ιρλανδικής Προεδρίας, η ατζέντα της, ε, η στρατηγική της ε, ασφάλειας για την ανάπτυξη. Αυτό που τονίζουμε είναι ότι ένα ασφαλές σταθερό οικονομικό περιβάλλον προωθεί τις οικονομικές δραστηριότητες, αναπτύσσει την εμπιστοσύνη στις επενδύσεις και βοηθά την νόμιμη οικονομία να αντισταθεί στις προσπάθειες της παραοικονομίας, να δυσδύσει σε αυτή, να υπάρχει ποινομοποίηση παρανομών εσόδων και η ακόλουθη έλλειψη εμπιστοσύνη, η άτυπη συνεδρίαση του Υπουργείου ΔΕΗ ε, στο Δουβλίνο ε, ασχολήθηκε με ένα κείμενο ακριβώς για αυτό το θέμα και ε, ότι τα κράτη-μέλη και οι υπουργοί θα δεσμευτούν για την όλη διαδικασία και μπορεί να δουν μία αναγκαιότητα σήμερα να διασφαλίσουν ότι τίποτα δεν θα μπει στο δρόμο, ότι να αναπτυχθεί όπως πρέπει η νόμιμη οικονομία. Και όπως σας είπα, αυτό ήταν από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην Ιρλανδική Προεδρία. Να αναφέρω επίσης εν συντομία το εξή η εμπρογνωμοσύνη της Europol ε, στο προσδιορισμό των εγκληματικών φαινομένων ε, είναι πραγματικά πρωτοπόρος από τη σκοπιά της Κόζη. Εμείς ε, θέλουμε να πάρουμε τη σόκτα και να αναπτύξουμε μια σειρά προτεραιοτήτων για δράση που ελπίζουμε να θετήσει ως συμπεράσματα το Συμβούλιο ΔΕΗ. Και στη συνέχεια θέλουμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά, να δράσουμε αποτελεσματικά σε αυτό το τομέα για να αναχαιτήσουμε αυτά τα φαινόμενα και να διώξουμε τους δράστες. Επίσης, ο ρόλος της ΚΟΖΗ είναι να διασφαλίσει ότι αυτά τα σχέδια είναι αποτελεσματικά, λειτουργούν σωστά και ότι τελικά έχουμε το μέγιστο όφελος από αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η Κομισιόν θα ήθελε να πει κάτι για τη συζήτηση αυτή. Παρακαλώ, κυρία Μίτση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Η Κομισιόν καλωσορίζει αυτή την σόκτα που όπως αναφέρθηκε μελετά τον κύκλο πολιτικής που θα μας συνοδεύσει τα επόμενα χρόνια. Επίσης θέλω να γνωρίσω την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει για την εκπόνηση αυτού του εγγράφου από τη Europol. Στο πλαίσιο της διαδικασίας του κύκλου πολιτικής θα ήθελα να αναφέρω ότι η Κομισιόν επικεντρώνεται σε ένα από τα στάδια που πρόκειται να λάβει χώρα και όπως ε, ανέφερε και ο κύριος ε, Πάουερ, η εκπόνηση μαζί με την Προεδρία του Συμβουλευτικού Εγγράφου που έχει σχεδιαστεί να καθοδηγήσει το Συμβούλιο ΔΕΗ στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για τον επόμενο κύκλο. Επίσης, είναι σημαντικό για την Κομισιόν να διασφαλίσει ότι υπάρχουν συνέργειε μεταξύ αυτού του κύκλου πολιτική και των προσανατολισμών της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πρωτοβουλειών. Και εγώ θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά στο θέμα της απειλής των πυροβόλων όπλων. Η ΣΟΚΤΑ επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε, ότι τα πυροβόλα έπλα είναι ο κοινό παρανομαστή σε όλα τα είδη σοβαρού και οργανωμένου κλίματο θα πρέπει να προσθέσουμε τα πυροβόλα έπλα που παρασκευάζονται και είναι αντικείμενο παράνομη εμπορία διασυνοριακά θέτουν άμεση απειλή στους Ευρωπαίους για τους Ευρωπαίους πολίτες και πολύ συχνά έχουν καταστροφικά αποτελέσματα όπως είδαμε στους πρόσφατους πυροβολισμούς στο Βέλγιο, στην Ορβηγία, στη Γαλλία. Επομένως, αυτοί οι καταστροφικοί προβολισμοί προκαλούν ανασφάλεια και όπως ξέρουμε προσελκύουν και την προσοχή του κοινού σε αντίθεση με τα ναρκωτικά ή τα παραποιημένα αγαθά που μπορούν να περιτελούν μία απειλή απέναντι στον καταναλωτή, τα πυροβόλα όπλα μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Και τα κράτη-μέλη επίσης έχουν ε, αναγνωρίσει κάτι τέτοιο και το Δεκέμβριο του 2010 τα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπογράμμισαν την ανάγκη για να υπάρχει βρεχπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη δράση κατά των βαριών πυροβολών όπλων και κατά της εμπορίας των όπλων εν αέρια. Έτσι λοιπόν ε, μας εκπλήσει ότι η ΣΟΚΤΑ δεν κάνει το βήμα του να συμπεριλάβει τα όπλα αυτά μεταξύ των κυρίων συστάσεων. Εμείς θα θέλαμε να δούμε να αντικατοπτρίζεται κάτι τέτοιο στις μελλοντικέ προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος. Καλωσορίζουμε την σημερινή συζήτηση την ευκαιρία που έχουμε για να έχουμε μια πολιτική συζήτηση για αυτόν τον κύκλο πολιτική και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ακούσαμε τα με, την άποψη των μελών αυτή τη Επιτροπή. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο στην ημερησία διάταξη εδώ. Και καθώς είμαστε και στα πλαίσια τα χρονικά, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Το οποίο είναι τροποποίηση τη απόφαση 2009, κάτω 935, ΔΕΗ, αναφορικά με τον κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με το οποίο η Europol συνάπτει συμφωνίε. Εισηγητή είναι ο κ. Κλέη. Σήμερα θα έχουμε παρουσίαση της πρότασης αυτής από τον Μαχώνη, ο οποίος είναι επικεφαλής του Διαχειριστικού Συμβουλίου της Europol και από τον κύριο Wainwright. Μόλις λοιπόν γίνει η αλλαγή εδώ στο βήμα, θα προχωρήσουμε. Παρακαλώ κύριο Μαχώνη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, θέλω από τη θέση μου να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε στην Επιτροπή σας σε σχέση με τις προτάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου προς το Συμβούλιο της Ένωσης για τις οργανώσεις με τις οποίες θέλει να συνάψει σχέση η Ευρωπόλ. Επειδή είναι πρώτη φορά που έρχομαι στην Επιτροπή σας, θα έπρεπε να σας πω λίγα για το ιστορικό μου. Είμαι αστυνομικός στην Ιρλανδική Γκάρντα τα τελευταία 26 χρόνια. Έχω μεγάλη εμπειρία αστυνομικής δράσης μεταξύ άλλων και την διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εγκληματιών. Τελευταία, από τη θέση μου έχω και διασυνδέσεις με την Ευρωπόλ και την Ιντερπόλ. Σήμερα με τον κύριο Ρόμπουιν θα σας δώσουμε μερικές πληροφορίες ανάλογα με το τι θα ζητήσετε. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπόλ, όπως ξέρετε, έχει εφαρμόσει συμφωνίες με 18 τρίτες χώρες και 13 διεθνείς οργανώσεις που βοήθησαν την Ευρωπόλ στην καταπολέμηση κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και ενεργειών στην Ένωση. Η πρόταση που έχετε μπροστά σας είναι μια σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου μας στις 3 και 4 Οκτωβρίου του 2012 για να προσθεθούν τέσσερις χώρες η Βραζιλία, η Γεωργία, το Μεξικό και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την εποχή που έγινε η σύστασή μας προς το Συμβούλιο ήμουν εκπρόσωπος της Ιρλανδίας, εκεί δεν ήμουν στη θέση που βρίσκομαι τώρα. Η ανάγκη να συναυθούν συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και οργανώσεις ε, προκύπτει από την ανάγκη πιο αποτελεσματικής καταπολέμησης της θερμοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και αυτό το έχουμε πλήρως αναγνωρίσει. Ως προς τη σύσταση, ο κατάλογος των χωρών και οργανώσεων με τον οποίο θέλουμε να συνάψουμε συμφωνία συζητήθηκε στην συνεδρίασή μας της 4ης Δεκεμβρίου του 2011 και τότε είχαμε καλέσει την Ευρωπόλ να μας εκφράσει τις ανάγκες της και τα ωφέλη και τα αρνητικά σημεία αλλαγής του καταλόγου της απαρίθμησης των χωρών με τις οποίες έπρεπε να συνάψουμε συμφωνίες. Η Γεωργία είχε ζητήσει να συμπεριληφθεί. Επομένως, μετά 1 και 2 Φεβρουαρίου του 2012 ο Διευθυντής της Ευρωπόλη επέβαλε ένα έγγραφο όπου εμφαίνονταν έξι χώρες και δύο οργανώσεις με τις οποίες είχε ενδιαφερόταν να συνάψει συμφωνίες η Ευρωπόλ. Σε εκείνη τη φάση μιλούσαμε για Βραζιλία, Μεξικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Γεωργία, Ιαπωνία και Νέα Ζηλανδία. Και οι οργανώσεις ήταν η Παγκόσμια Τράπεζα, και το ΣΕΛΕΚ. Γνωρίζαμε τις πολιτικές προτεραιότητες, αλλά ο κατάλογος αυτός βασιζόταν μόνο και μόνο στα ενδιαφέροντα της Ευρωπόλου. Και καλέσαμε λοιπόν τον Διευθυντή να ζητήσει από τη Βραζιλία, το Μεξικό και τη Νέα Ζηλανδία να προσέλθουν στην επόμενη συνεδρίαση για να παρουσιάσουν την περίπτωσή τους. Εις 7 Ιουνίου 2012 ο Διευθυντής υπέβαλε εκθέσεις για τη Βραζιλία, τη Γεωργία και το Μεξικό και κατέληξε ότι ήταν μεγάλη προτεραιότητα η σύναψη συμφωνίας με τις δύο πρώτες στο Μεξικό, επίσης θεωρήθηκε σημαντικό. Με βάση τις υποβολές που έγιναν, περιγράφτηκαν και οι κυρίες εγκληματικέ δραστηριότητες που δικαιολογούν την προσθήκη των χωρών αυτών στον κατάλογο για τη Γεωργία. Λεωφορηθήκαμε ότι στη Γεωργία το οργανωμένο έγκλημα αυξάνεται και δρά και στην Ένωση. Πολλές χώρες μέλη έχουν προβλήματα από γεωργιανές εγκληματικές ομάδες. Μία συμφωνία συνεργασίας με τη Γεωργία θα επέτρεπε την ανταλλαγή πληροφοριών και αναλύσεων και θα βοηθούσε την Ευρωπόλ να έχει μια καλύτερη στρατηγική έποψη για το γεωργιανό οργανωμένο έγκλημα στην Ένωση. Επίσης θα βοηθούσε αυτό την Ευρωπόλ να είναι σε ισχυρότερη θέση για να αντιμετωπίσει έρευνες που αφορούν χώρες μέλη που έχουν σχέση με γεωργιανά εγκλήματα με εγκλήματα γεωργιανών οργανώσεων. 11 ε, ο γεωργιανό οργανωμένο έγκλημα θεωρήθηκε σαν κάτι πολύ σημαντικό για τις κλοπές και διαρρήξεις. Η βάση του βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ευρωπόλ σε μία έκθεσή της για το έγκλημα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη θέλησε να ασχοληθεί και με γεωργιανές εγκληματικές ομάδες που δρούν μέσα στην Ένωση για κλοπές και διαρρήξεις, παράνομη μετανάστευση, απάτες και απομιμήσεις, ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος και ελευθερμπορία ναρκωτικών. Και κατέληξε ότι αποτελεί απειλή το γεωργιανό οργανωμένο έγκλημα στο εσωτερικό της Ένωσης και απαιτείται ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Ευρωπόλ και Γεωργίας. Για τη Βραζιλία τώρα. Η έκθεση αυτή έλεγε ότι το κοινό σχέδιο Βραζιλίας Ένωσης που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2011 στη Βραζιλία ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βραζιλία να συνεργαστούν για την πρόληψη και αντιμετώπιση της κατάχρησης των δημοσιονομικών του συστημάτων για το ξέπλυμα προμήκου χρήματος και προέβλεπε την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και πληροφοριών για την καλύτερη δίωξη των εγκλημάτων και την βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας των. Ως προς τις ε, σχέσεις Ευρωπόλ και συγκεκριμένων κρατών για αντιμετώπιση βραζιλιανών εγκλημάτων σημειώσαμε ότι επειδή πολλοί Ευρωπαίοι μεταναστεύουν στη Βραζιλία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την αυξημένη δραστηριότητα βραζιλιανών εγκληματικών ομάδων που έρχονται στην Ευρώπη μέσω της παράνομης μετανάστευσης. Το 2011 το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιούσε και Λατινοαμερικανούς για δουλεμπορία. Εκτός αυτού χρήματα από το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών στη Νότια Αμερική έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται και στο εμπόριο ειδών ζώων που βρίσκονται υπό εξαφάνιση. Επομένως χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία και για τη Βραζιλία στους εξής τομείς. Εγκλήματα στον τόπο εργασίας, απομιμήσει σε ευρώ, πλαστά ευρώ και το 14 σημειώνουμε ότι θα γίνει το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στη Βραζιλία και έτσι θα δοθούν πρόσθετες ευκαιρίες για το οργανωμένο έγκλημα. Και η έκθεση επίσης αυτή ζητούσε περισσότερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπόλ και Βραζιλίας. Το Μεξικό τώρα. Αυτή η έκθεση έλεγε ότι υπάρχει προς στιγμήν χαμηλή δραστηριότητα, χαμηλές, χαμηλό επίπεδο σχέσεων μεταξύ Ένωσης Ευρωπόλ και Μεξικού. Αλλά έλεγε επίσης ότι οι απειλές προς την, Ευρωπαϊκή, προς την εσωτερική ασφάλεια της ε, Ένωσης ενδιαφέρουν τους εξής τομείς για το Μεξικό εγκλήματα εργασίας, γιατί ακούσαμε και πριν να λέγεται ότι υπάρχει νέα απειλή από μεξικανικά καρτέλ στον τομέα της λαθεμπορίας ναρκωτικών. Παραδοσιακά οι Μεξικανοί περιορίζονται στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, και ο κύριος προμηθευτής τους είναι η Κολομβία εδώ. Αλλά τώρα, πρόσφατα, έχουν υπάρξει και κατασχέσεις ναρκωτικών που δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εμπορία και από το Μεξικό προς την Ευρώπη. Παράγει μεταμφεταμίνη και μεγάλε ποσότητες κοκαίνης 400 κιλά κατασχέθηκαν στην Ισπανία πρόσφατα με προέλευση Μεξικό. Και το δουλεμπόριο και εμπορία ανθρωπίνων όντων, ιδίω ανατολικοευρωπαίων γυναικών από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έχουν μεταφερθεί στο Μεξικό. Τρομοκρατία. Έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν τρομοκρατικές οργανώσεις στο Μεξικό που διενεργούν απάτες με πιστοτικές κάρτες στην Ευρώπη και προέρχονται από το Μεξικό. Και μερικές είναι οργανωμένες με μοτοσικλέτες και μοτοσακό. Επίσης υπάρχει αυξημένη τάση δραστηριότητα των εγκληματικών οργανώσεων του Μεξικού στην Ευρώπη, αλλά η Ευρωπόλ δεν έχει ακόμη αρκετά στοιχεία για να το αποδείξει, αλλά και οι ενδείξεις που έχουμε είναι αρκετά σοβαρές ώστε να δοθεί προτεραιότητα στη συνεργασία με το Μεξικό. Στην ίδια συνεδρίαση 6-7 Ιουνίου ο Διευθυντής συνέστησε οι τρεις αυτές χώρες να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα στον κατάλογο των χώρων με τις οποίες θέλουμε να συνάψουμε σχέσεις και τον, η Κομισιόν τόνισε ότι οι επόμενες συμφωνίες θα συναυθούν με διαφορετικό πλαίσιο και θα δοθεί μεγάλη προτεραιότητα στη Γεωργία, στο θέμα των θεωρήσεων και στη συμφωνία με το Μεξικό. Πολλά μέλη του Συμβουλίου μας θεωρούσαν ότι ότι η Ευρωπόλ πρέπει να περιοριστεί στις βασικές της δραστηριότητες και να μην εγκρίνει περαιτέρω ανάπτυξή τους. Τελικά η Γερμανία πρότεινε η Ευρωπόλ να προετοιμάσει μια έκθεση για συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό το υποστήριξαν και άλλες χώρες μέλη και συμφωνήθηκε το Συμβούλιο να καλέσει την Ευρωπόλ να κάνει μια έκθεση για συμφωνία συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που να εξεταστεί από το Συμβούλιο. Υπευλήθη γραπτό στις 25 Ιουνίου και μέχρι τις 6 Ιουλίου το εξέτασε. Τελικά όμως υπήρξε αρνητική γνωμοδότηση για σύναψη σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυρέτα με επιστολή της Επιτροπής της 9 Ιουλίου και ζητήθηκε νέα συζήτηση της περίπτωσης των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπόλ για χώρες εκτός των τριών που είχαν εγκριθεί ήδη. Στην έκθεση που γράφτηκε από το Συμβούλιο τονίζονταν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ε, πρέπει να ενδιαφέρουν όλο και περισσότερο την Ένωση ως προς την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος γιατί έχουν γίνει κέντρο δημοσιονομικού εγκλήματος και έχουν ταυτιστεί ως κέντρο ξεπλήματος βρωμίκου χρήματος και διαφόρων απατών καθώς και απατών ως προς το ΦΠΑ γιατί πρόκειται για μία χώρα ελευθέρων συναλλαγών που έχει πρόσβαση στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές και επομένως στο λαθρεμπόριο σιγαρέτων. Για το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι διαμετακομιστικός κόμβος και για ναρκωτικά και για άλλα εμπορεύματα. Και μεγάλο ποσό χρημάτων επενδύεται από τα Αραβικά Εμμυράτα στο λαθρεμπόριο στην Ευρώπη. 6 εκατομμύρια ευρώ σε κατασχέσεις από λαθρεμπόριο από τα Αραβικά Εμμυράτα. Σημαίνουν ότι η Ευρωπόλ είναι σημαντικός παράγοντας στην καταπολέμηση και του λαθρεμπόριου. Λόγω δε της αυξανόμενης σημασίας των Ηνωμένων Αραβικών ως κέντρο διαμεκομιστικών απατών, η έκθεση για, τα, για αυτά έλεγε ότι υπάρχει λόγος για σύναψη συμφωνίας Ευρωπόλ Αραβικών Εμμυράτων στις 4 Οκτωβρίου ξανασυζητήθηκε το θέμα και το Συμβούλιο συμφώνησε να συσταθεί να συμπεριληφθούν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στον κατάλογο των χώρων Στις 4 Οκτωβρίου του 12 ο προκάτοχός μου πληροφόρησε τη Γενική μας Γραμματεία για τις συστάσεις του Συμβουλίου να συμπεριληφθούν οι τέσσερις πλέον αυτές χώρες στις πρωτεύουσε για συμφωνία. Και κατέθεσε στη Γενική Γραμματεία όλες τις εκθέσεις που σας ανέφερα προηγουμένως. Το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε να στα επόμενα χρόνια σύντομα να εφαρμοστούν όλα αυτά και οι συμφωνίε συνεργασία. Παρόλα αυτά, η σύσταση του Διοικητικού Συμβολίου βασιζόταν μόνο στι επιχειρηματιακέ ανάγκε τη Ευρωπόλ και όχι σε γενικότερε πολιτικέ προτεραιότητε. Και η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθετική διαδικασία του άρθρου 26α επειδή η εγκληματικότητα αυξάνει και αυξάνεται διεθνώ, η συνεργασία πρέπει να είναι αποτελεσματική και διεθνή. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ευρωπόλ πρέπει να διασφαλίσει ότι θα ληφθούν έγκαιρε αποφάσει για να μπορεί η Ευρωπόλ να, κάνει, να ενεργήσει την ισχυρότερη δυνατή συνεργασία. Η ευθύνη τη Ευρωπόλ καθώ και του διαχειριστικού του διοικητικού τη Συμβουλίου είναι να αυξήσει την ασφάλεια όλων των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό Καλό την Επιτροπή σας να δεχτεί τη σύστασή μας προς το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Θα θέλετε και εσείς, Wainwright, να πείτε δύο λόγια. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ομάνου έχει καλύψει πολλές λεπτομέρειες. Θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσω και λίγα λεπτά για να εξηγήσω κάποια από τα ζητήματα που ανάφερε. Καταρχάς, η εξωτερική ατζέντα της Europol είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντική. Δεδομένη της παγκοσμιοποίηση του οργανωμένου εγκλήματο, προφανώς χρειάζεται ισχυρή στρατηγική προ τα έξω. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλο και πιο πολύ. Και ο εισηγητής από την Επιτροπή ΚΡΙΜ καλεί τι υπηρεσίε να σφίξουν σχέσεις με τους ευρωπαϊκούς εταίρους. Ακολουθούμε μια διαδικασία η οποία ορίζεται στο πλαίσιό μας και μια λίστα που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει επί της ουσίας μια μελέτη των προτύπων προστασίας δεδομένων στις τρίτες χώρες. Ανεξάρτητη αξιολόγηση από τη σχετική υπηρεσία πρωτού συνάψουμε την σύμβαση και μετά ε, αυτό εξετάζεται στο Συμβούλιο. 25 χώρες στην παρούσα φάση στον κατάλογο. Καμία δεν έχει πλήρη ε, συμφωνία για πλήρη ανταλλαγή. Όχι, συγγνώμη. Ε, έχουν 25 χώρες τέτοια δικαιώματα ανταλλαγής δεδομένων, ενώ εννέα άλλες δεν έχουν τέτοια δικαιώματα. Η λίστα όμως είναι δυναμική και αλλάζει ο κόσμος του εγκλήματος, όπως ε, αναφέραμε και στις 8, και εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε, όπως είπε ο Πρόεδρος. Ο κατάλογος τροποποιήθηκε το 2009 για τελευταία φορά και πολλά έχουν συμβεί ε, τότε όπως αναγνωρίζει και η ΣΟΚΤΑ. Και γι' αυτό Η Ευρωπόλ έχει εντοπίσει τις τέσσερις χώρες αυτές όπου το λειτουργικό ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσαμε για την αύξηση των μεξικανικών καρτέλ ναρκωτικών και πώς έχει καταστεί, για παράδειγμα, μεγάλη πλατφόρμα για απάτη σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ. Αναγνωρίζω ότι θα λάβουμε και την ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα κανονισμό της Ευρωπόλης. Ίσως θα είναι πιο απλό να περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία το ξεκινήσουμε εμείς μια, παράλληλα, μια παράλληλη νομοθετική διαδικασία και καταλαβαίνω ότι οι καταστάσεις είναι πέρα, απέχουν παρασάγκασα από το να είναι ιδανικέ. Αλλά μπορεί να έχουμε περιμένει τέσσερα χρόνια για να προσαρμόσουμε τη λίστα Πόσα άλλα χρόνια θα χρειαστεί να περιμένουμε προτού εφαρμοστεί ο κανονισμός της Europol. Πρόκειται για μια σκέψη απλά που αποτυπώνει τις σκέψεις της Europol για την ε, τρέχουσα κατάσταση στο οργανωμένο έγκλημα και πώς ε, πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς αναλόγως. Και εδώ κλείνω. Αυτό που δεν αποφασίζουμε με την πρόταση αυτή είναι να ολοκληρώσουμε τις συμφωνίες με τις χώρες αυτές. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης διαδικασίας. Ανοίγουμε απλά μία πόρτα και μετά από αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα θέματα προστασίας δεδομένων. Δεν υπάρχει κανένας αυτοματισμός από, το, από τη στιγμή που θα μπουν στην λίστα του Συμβουλίου και ε, μια ενδεχόμενη σύναψη σύμβαση. Απλά ανοίγει η πόρτα για μια ενδεχόμενη συμφωνία και αυτό το χρειάζεται η Europol για να μπορέσει να διατηρήσει την αποτελεσματικότητά τη ό,τι αφορά την υποστήριξη των χωρών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε τώρα τρία άτομα που έχουν στήσει το λόγο. Καταρχήν ο κ. Κλέη, κατόπιν η κυρία Ματιέ και ο τελευταίο ομιλητή. Κ. Κλέη, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά ε, να ευχαριστήσω τον κύριο Μαούν και την, ε, τον κύριο Ράιτ για την πολύ εκτενή παρουσίασή τους. Το ερώτημα τώρα που ανακύπτει προκύπτει από το λειτουργικό σκέλος της Ευρωπόλ και από κάποια κράτη-μέλη και αναφέρεται Ja, dus op een aantal zaken die operationeel zijn αναφέρεται σε κάποια λειτουργικά στοιχεία. Καλό θα ήταν λοιπόν σε κάθε περίπτωση να διαθέτουμε τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, μάλλον που μας παρουσιάστηκαν, ιδιαίτερα τις πληροφορίες του κ. Μαούνη, να τις έχουμε και σε γραπτή μορφή στη διάθεση της Επιτροπής μας, προκειμένου να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι θα είχαμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στο ερώτημα του ποιοι είναι οι λειτουργικοί λόγοι για, την, για τη συμπερίληψη και άλλων χωρών στην λίστα αυτή. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες άλλες, αλλά υποθέτω ότι πρόκειται για σύναψη συμφωνιών που είναι και λειτουργικές. Με ανταλλαγή δηλαδή προσωπικών δεδομένων. Μία άλλη ερώτηση, η ερώτηση που έχει να κάνει με τη χρονική συγκυρία. Υπάρχει και άλλη λίστα τρίων των χωρών με τις οποίες γίνονται διαπραγματεύσεις και με τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις ακόμα. Η Κίνα, η Ινδία, σημαντικές χώρες, το Μαρόκο, το Ισραήλ. Και σε τι βαθμό η Ευρωπόλ έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες αυτές και παράλληλα και με τις άλλες τέσσερις χώρες Πώς λειτουργεί κάτι τέτοιο σε πρακτικούς όρους. Ή μήπω οι διαπραγματεύσει με την Κίνα, την Ινδία, το Μαρακό και την Ισραήλ έχουν σταματηθεί, έχουν παγώσει προσωρινά. Και πότε θα ήθελε η Ευρωπόλη να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την Γεωργία, τα Αραβικά Εμμυράτα, τη Βραζιλία και το Μεξικό. Ο κύριος ε, Wainwright απάντησε ήδη στο ερώτημα το οποίο μοιραία προκύπτει, τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις και πότε μπορούμε να ελπίζουμε σε έναν καινούριο κανονισμό σε ό,τι αφορά την τη της Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ματιού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απριόρι είμαστε αρκετά θετικοί απέναντι σε αυτή τη συμφωνία εταιρική σχέση, δεδομένου τη ευαισθησία αυτών των χωρών, αλλά έχω την ίδια ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα. Εσεί αναφερθήκατε ναι, σε αυτό, αλλά θα ήθελα να μου πείτε κάποιε λεπτομέρειε για το θέμα αυτό και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αναφερθήκατε σε αυτό το ζήτημα και το έκανε και ο συγητής. η κυρία Χιμένες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Διευθυντή της Europol και τον κύριο Μαχώνη. Θα ήθελα να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση για το Μεξικό. Γιατί τη δική μου αντιπροσωπεία είχε τη δυνατότητα να μεταβεί πολλές φορές στο Μεξικό και συναντηθήκαμε με τον Υπουργό εσωτερικών και με άλλου ε, υπεύθυνου για την καταπολεμήση του οργανωμένου εγκλήματο. και έχουμε προγραμματίσει και το Μάιο ένα ταξίδι όπου θα συζητήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο ναρκωτικών. Και φυσικά πάντοτε συζητάμε και το θέμα της συνεργασίας με την Europol. Θέλω να ρωτήσω, πώς πιστεύετε εσείς ότι εμείς οι βουλευτές μπορούμε να συνεργαστούμε και να βοηθήσουμε, να προωθήσουμε αυτές τις συμφωνίες μεταξύ Μεξικού και Ευρωπόλ, στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Μεξικό-Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίση, θα ήθελα να μου πείτε αν σήμερα υπάρχει κάποιο είδου συμφωνίας μεταξύ Ευρωπόλ και Μεξικού και αν από το Μεξικό υπάρχει βούληση συνεργασίας, αν αυτοί πράγματι ενδιαφέρονται για τις συμφωνίες αυτές. Επίσης, μίλησατε για εμπορία ανθρώπων, για εμπορία ναρκωτικών, αλλά και για τρομοκρατικές ομάδες στο Μεξικό και θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς σε τι, αναφερθεί, σε τι αναφερόταν αυτό. Πρόεδρος, σε ευχαριστώ. Πριν να δώσω στο λόγο καταρχήν στον κύριο Μαχωνή και κατόπιν στον κύριο Ράιτ να κάνω κι εγώ μία σύντομη ερώτηση για τη Γεωργία. Νομίζω ότι οι εγκληματικές οργανώσεις ε, στη Ρωσία συνήθως έχουν μία εθνική βάση και όταν ε, μιλάτε για την αντιμετώπιση του γεωργιανού εγκλήματος, μάλλον αυτό συνδέεται και με την καταπληρωμή του ρωσικού εγκλήματος. Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την Σκοπιά και σε σχέση με τις ερωτήσεις που τέθηκαν, θα ήθελα να σας πω ότι θα σας διαβιβάσω ένα αντίγραφο της παρουσίασής μου και θα βεβαιωθώ ότι θα το λάβετε ως εκπρόσωπος των κρατών μελών και πρόεδρος του Συμβουλίου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε και κατόπιν να υποστηρίξουμε τη Europol. Στον αναπτύξει συνεργασία με τρίτες χώρες. των οποίων ε, η εγκληματικότητα έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και στους μεμονωμένους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι συζητήσεις που ξεκίνησαν το 2011 και ολοκληρώθηκαν με την απόφαση τον Οκτώβριο του 2012 έγιναν καθαρά σε επιχειρησιακή βάση. Και υποθέτω με την εμπειρία των αρχών επιβολής του νόμου που υπάρχει, υποθέτω ότι η ρευστότητα του οργανωμένου κλίματος ε, και ε, οι διάφορες εξελίξεις, οι αλλαγές που συμβαίνουν καθημερινά, θέτουν νέες προκλήσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε εμείς σε θέση να αναπτύσσουμε, να εξελισσόμαστε γιατί αυτές οι συμφωνίες αργούν να ολοκληρωθούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί έλεγχοι και διασταυρούμενοι έλεγχοι και από τα δύο μέρη για να διασφαλίζεται ότι τα πρότυπα που εμείς ε, θέλουμε να τηρούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν και στις άλλες χώρες, κυρίως ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων. Επομένως, οι αποφάσεις που λαμβάνονται για να συνεχίσει η Europol τη σύνέψη αυτών συμφωνιών είναι ότι θα πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει όταν θα ισχύσει ο νέος κανονισμός και τότε όταν θα ισχύσει ο νέος κανονισμός θα μας πει πώς τελικά θα σφραγιστούν αυτές οι συμφωνίες, αν τελικά σφραγιστούν. Νομίζω ότι αναφέρθηκα στο όσο το ναι, και ξέρω ότι η Γεωργία θέλει να μπει στη διαπραγματεύση. έχει εκφράσει τον ενδιαφέρον αυτό σε αρκετά κρατημέλη και θα ήθελα να συνεργαστεί βέβαια σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Φυσικά το οργανωμένο έγκλημα από τη Γεωργία έχει αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. αλλά ε, υπάρχει και συνεργασία και με όμορες χώρες. Και το έχουμε αυτό δει τακτικά. Έχουμε σχετικές εμπειρίες σε κράτη-μέλη. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ο κύριος Wainwright. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Κλέης, και τους υπόλοιπους σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις αυτές. Εμείς συνηθίζαμε να έχουμε παράλληλες ε, συζητήσεις γιατί μπορεί να χρειαστεί τέσσερα χρόνια να ολοκληρωθεί μια συμφωνία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μία να διαδέχεται την άλλη. Επομένω. είμαστε συνηθισμένοι στο να υλοποιούμε διάφορε διαπραγματεύσει σε διάφορα στάδια. Αυτή τη στιγμή τα πάμε αρκετά καλά. Έχουμε ολοκληρώσει πρόσφατα μια σειρά διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και το Λιχτενστάιν που αντικατοπτρίζουν μέρη την επιθυμία μας να θέσουμε προτεραιότητα στη συμφωνία συνεργασίας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Υπάρχει και μια άλλη συμφωνία όπως αυτή με τη Ρωσία που είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση, ελπίζω να ολοκληρωθεί φέτος. Με το Ισραήλ υπάρχει μια καθυστέρηση, όμως ε, και εκεί έχουμε προχωρήσει σημαντικά μόνο μία πρόκειται να ξεκινήσει για τη Σερβία. Και έχουμε και άλλε διαπραγματεύσει που τον κατάλογο δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη καθόλου. Η Ινδία, παραδείγματο χάρη. Και αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονό ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και από την άλλη πλευρά φυσικά πριν ε, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Συνήθω ε, ισχύει αυτό όμω σε αυτέ χώρε προ στιγμή. Να έχουμε τι συζητήσει για το Μεξικό και για τη Βραζιλία. Υπάρχει υψηλή πολιτική βούληση που εκφράζεται συχνά σε υψηλό πολιτικό επίπεδο από τους πρεσβευτές αυτών των χωρών, στις Βρυξέλλες, παραδείγματο χάρη, από τους ε, αρχηγούς τη αστυνομία και στι δύο περιπτώσει, όμως δεν ε, αμφισβητώ ότι πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον ε, στην περίπτωση αυτή. Και επίσης βλέπουμε και ένα αυξανόμενο συνδεσμό οργανωμένων κλίματος μεταξύ διάφορων υπήρων και αναφέρουμε συγκεκριμένα στη διακίνηση ναρκωτικών. Η κυρία Ματιέ ρώτησε για τη διαδικασία εδώ. Όπως είπα νωρίτερα, εδώ ανοίγουμε τις πόρτες, είναι μακρά η διαδικασία. Σε οποιαδήποτε συμφωνία που τελικά θα, μετα... θα επιτρέψει τη διαβίβαση δεδομένων, για οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να μελετήσουμε τις ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας των δεδομένων σε εκείνη τη χώρα και φυσικά οι υπαλληλοί μας εξετάζουν και ελέγχουν την ομοθεσία, πώς τίθεται σε εφαρμογή, υλοποιούν μια έκθεση ανεξάρτητα και επίσης υποβάλλουν και μια έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κάνει μια σύσταση στο Συμβούλιο και μόνο τότε όταν έχουν υλοποιηθεί όλα αυτά τα βήματα μπορούμε να συνάψουμε τη συμφωνία. Πολύ συχνά βρίσκουμε προβλήματα καθ' όλη τη διαδικασία με τα πρότυπα προστασία των δεδομένων και μπορεί να χρειαστούμε και ακόμα δύο χρόνια για να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα εμπόδια. Επομένω, δεν είναι εύκολη και αυτό με τη διαδικασία πάντοτε. Υπάρχει πραγματικό τεστ των πρότυπο προστασία των δεδομένων πριν να μπορέσει να ολοκληρωθεί, να συναυθεί μια συμφωνία. Αυτή είναι η διαδικασία που ισχύει σήμερα και πιστεύω ότι και στην περίπτωση αυτή μπορούμε να την εφαρμόσουμε και να έχουμε τους απαραίτητους πόρους να διαπραγματευτούμε αυτές τις συμφωνίες με τον κανονικό τρόπο. Ευχαριστώ κύριοι. Εδώ ολοκληρώνουμε και το σημείο 14 παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα εκ νέου να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους ε, της ε, Europol θα ήταν ενδιαφέρον όμως να ακούσουμε και την άποψη του Συμβουλίου και του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν για τα θέματα αυτά. Okay. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτοιμη είναι η εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή εξάφρασε τις απόψεις της όπως αναφέρθηκε και σε αυτό ο κ. Μακόνη, σε διάφορες συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ε, Europol σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την συμπερίληψη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον κατάλογο εν δυνάμει καινούριων εταίρων της Europol. Η θέση η οποία εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να φανεί και μέσα σε μια επιστολή που απέστειλε η Επίτροπος Μάλμστρομ στους υπηρεσίες των ιστορικών υποθέσεων τον προηγούμενο Ιούνιο, όπου και σύστησε προσοχή σε ό,τι αφορά τη σύναψη συμφωνίας με τρίτες χώρες, δεδομένου αφενός ότι είναι πολύ ιδιαίτερη η κατάσταση δημοσιονομική και την είναι πολύ πόρη. Αυτό επηρεάζει τους πάντες και τις υπηρεσίες και ασφαλώς ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να θέσουμε σωστές προτεραιότητες. Και αφετέρου του γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν συμφωνίες με τρίτες χώρες όπου υπάρχει γεωγραφικό συμφέρον αλλά και θεματικές προτεραιότητες στον τομέα των ιστορικών υποθέσεων. Και το τελευταίο αυτό ζήτημα καλύπτει και, την Ευρωπαϊκή, και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και του στρατηγικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Αραβικά Εμμυράτα δεν υπάγονται σε καμία από τις δύο αυτές κατηγορίες. Πιο γενικά, ε, όπως αναφέρθηκε και από μια σειρά ομιλητών, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας, η Europol, και αναφέρομαι στον κανονισμό που θα εγκριθεί για το Europol, το τρέχον καθεστώς που βασίζεται στις εφιστάμενες αποφάσεις για την Europol σταδιακά θα καταργηθεί και η διαδικασία που επιτρέπει στην Europol να συνάπτει η ίδια συμβάσεις ε, με τρίτες χώρες στον τομέα της ασφάλειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, να μας στείλετε, αν θέλετε, ένα αντίγραφο της επιστολής αυτής, γιατί κατά τη διάρκεια της συζήτηση για το Συμβούλιο του Πολιετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ακολουθήθηκε μία, θεωρώ, ανόητη προσέγγιση. Και βλέπουμε ότι με την προσέγγιση αυτή τώρα δεν έχουμε επαρκείς πόρου και θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή πώ πανώνται αυτοί οι πόροι. Θα ήθελα λοιπόν να έχω αυτή την επιστολή, αν θέλετε. Please. Χωρίς μικρόφωνο μιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπρόσωπο την Προεδρία. Για το θέμα αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει την απόφαση με σαφήνεια και ο διευθυντή ε, τη Europol ε, τόνισε τι και απαιτήσει ε, και η ομάδα εργασία επιβολή του νόμου υιοθέτησε τη στάση του Διοικητικού Συμβουλίου και τώρα αναμένουμε τη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προωθηθεί η απόφαση για υιοθέτηση. Όμω η Προεδρία υποστηρίζει την απόφαση αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο. Τώρα έχουμε το σημείο 15, τα διάφορα. Δεν υπάρχει κάτι. Σημείο 16, επόμενη συνεδρίαση στις 8 Απριλίου στις 3 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ.